Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Καλώς ήλθατε στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού, η οποία έχει μια αρκετά α, επιβαρημένη ημερησία διάταξη. Ο κύριος Ότης ζήτησε να τροποποιηθεί, η κυρία μάλλον, συγγνώμη, με συγχωρείτε, η κυρία Ότης ζήτησε να τροποποιηθεί η σειρά της ψυχοφορίας, γιατί έχει να προλάβει ένα, μια πτήση. Αν δεν υπάρχει πρόβλημα, τότε να γίνει. Επισημαίνω ότι η συνεδρίασή μας είναι ε, δημοσία και επομένως μεταδίδεται και από το διαδίκτυο και αυτό το βρίσκουμε ιδιαίτερα ικανοποιητικό και επισημαίνω επίσης ότι στα πλαίσια της κινητοποίησης των συνεργατών μας, job rotation, έχουμε νέο συνεργάτη στη γραμματεία, Φίλιπ Γκότς, που αποτελεί πλέον μέλος της γραμματείας μας. Καλώς ήλθατε. Ε, είχα ήδη την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί σας το ανακοινώνω ωστόσο και στην σημερινή δημόσια συνεδρίαση. Θέμα 3 της ε, ημερησίας διατάξεως, προστασία των οικονομικών συμφερόντων των κοινοτήτων, καταπολέμηση της απάτης, αγώνας κατά της απάτης, πάντα σημαντικό, βέβαια και τώρα πια ιδιαίτερα επίκαιρο θέμα και επ' αυτού ε, απευθύνω το καλό ορίσατε στον Επίτροπο κύριο Σέμετα Ας ακούσουμε πρώτα την δική σας τοποθέτηση για να περάσουμε μετά στην συζήτηση. Και μετά θα ακούσουμε την παρουσίαση του κυρίου Κέσλερ, Διευθυντού της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Απάτης, Όλαφ. Καλώς ήρθατε κύριε Επίτροπε. Είστε πάντοτε καλόδεχτο στην Επιτροπή μας και χαιρόμαστε που ως Επίτροπος λαμβάνετε πολύ σοβαρά υπόψη σας το θέμα αυτό. Εμείς βεβαίως έχουμε καθήκον να ελέγχουμε το τι πράττει η Κομισιόν, αλλά ταυτόχρονα υποστηρίζουμε τα πρόσωπα εκείνα τα οποία εργάζονται για την προάσπιση των συμφερόντων της Ένωσης. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. τους δύο τελευταίους μήνες είναι σήμερα η δεύτερη φορά που έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας τις πολιτικές που ακολουθούμε για την προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Θα σας δώσω μια συνολικότερη επισκόπηση για το πώς κινήθηκε η κατάσταση το 2011. Έχουμε και την ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον αγώνα κατά της απάτης κατά ε, εφαρμογή του άρθρου 325 της Συνθήκης. Όπως κάθε χρόνο η έκθεση μας δίνει μια στατιστική επισκόπηση όλων των ε, ατασταλιών που έχουν σημειωθεί στις χώρες μέλη και τις οποίες αυτές έχουν ανακοινώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα δείτε τώρα ωστόσο ότι τώρα υπάρχει μια σαφής διάκριση μεταξύ ε, σταλιών οι οποίες οφείλονται σε απάτη και άλλες οι οποίες ανακοινώνονται ως μη προϊόν απάτης. Μόνον οι πρώτες, δηλαδή όσες έχουν δηλωθεί ως αποτέλεσμα απάτης, θεωρούνται απάτη. Δεύτερο, η έκθεση του 2011 εναρμονίζει τις πληροφορίες σχετικά με την ανάκτηση αδικαιολογήτως καταβληθισών πληρωμών και την εγγραφή τους στους ετήσιους λογαριασμούς, ώστε να αποφευθούν ορισμένες δυσχέρειες για την ε, αντιπαραβολή πληροφοριών σε έξι ετήσιους λογαριασμούς. Αυτό προέκυψε από την ε, επεξεργασία σχολείων που έλαβα από την Επιτροπή σας και με τα οποία συμφώνησα. Ελπίζω ότι θα βρείτε την φετινή ετήσια έκθεση πραγματικά χρήσιμη. Επίσης, και μετά από παλαιότερα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η έκθεση του 2011, όπως και οι προηγούμενες, περιλαμβάνουν έξτρα πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο θέμα, το οποίο φέτος είναι η έλεγχη για την καταπολέμηση της απάτης στο χώρο της πολιτικής συνοχής. Επίσης, το ψήφισμα του Κοινοβουλίου για το έτος 2011 μας έδωσε πολύ χρήσιμες ενδείξεις, τις οποίες λάβαμε υπόψη στην σύνταξη της έκθεσής μας και παρακολουθούμε την εξέλιξή τους. Η έκθεση συμπληρώνεται από τέσσερα έγγραφα εργασίας. Περιλαμβάνεται σε αυτά ένα νέο. Οι συμβολές των χωρών μελών για την εφαρμογή του άρθρου 325 της συνθήκης, η συνέχεια που δίνεται στις συστάσεις προηγουμένων εκθέσεων, η στατιστική αξιολόγηση των irregularities που έχουν ανακοινωθεί το 2011 και η νέα στοιχεία μεθοδολογίας για τη στατιστική αξιολόγηση των ε, ε, περιπτώσεων που μας υποβλήθηκαν για το 2011. Επί της ουσίας έχω τρία ε, σημαντικά στοιχεία εξελίξεων από την έκθεση του 2011. Πρώτα, βλέπουμε ότι τα συστήματα ε, διοίκησης και ελέγχου έχουν βελτιωθεί σημαντικά και αυτό απηχείται σε μια συνολική αύξηση στις ε, κοινοποιηθήσεις περιπτώσεις που μας υποβλήθηκαν. Αυτό βεβαίως έχει ληφθεί υπόψη και από το ελεγκτικό συνέδριο. Βλέπουμε εξάλλου από την φετινή έκθεση ότι έχει βελτιωθεί και η ανάκτηση στο έτος 2011. Τρίτο, ένας αριθμός πρωτοβουλειών πολιτικής που έχουν προωθηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ενισχυθεί ο αγώνας κατά της απάτης ακόμα περισσότερο. Επιτρέψτε μου τώρα να έρθω σε περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτά τα τρία σημεία. Η έκθεση δείχνει ότι ο αριθμός παρατυπιών που οφείλονται σε απάτη μειώθηκε κατά 35% σε σύγκριση με το 2011. Επίσης, το συνολικό ύψος μειώνεται κατά 37% και φτάνει στα 404 εκατομμύρια ευρώ φέτος. Ο αριθμός παρατυπιών που δεν κοινοποιήθηκαν ως δόλιες μειώθηκαν επίσης κατά 17%. Εκτιμόμενο ποσό μειώθηκε κατά 6% σε 1,5 δις ευρώ. Επίσης, εμείς δεν ισχυριζόμαστε ότι αυτές οι σημαντικές βελτιώσεις οφείλονται σε βελτίωση χρήσεων των ταμείων. Ένα μέρος από τι μειώσεις αυτές ήταν αναμενόμενο και είχε μάλιστα προβλεφθεί στην έκθεσή μας το 2010. Εγώ μιλώ για το μέρος εκείνο που συνδέεται με τον κυκλικό χαρακτήρα ορισμένων προγραμμάτων και ιδίως στον τομέα της πολιτικής συνοχής, όπου οι κοινοποιηθήσει παρατυπίες ε, μειώθηκαν σημαντικά κατά 45%. Λαμβάνοντας ακόμη υπόψη τον παράγοντα αυτών, Υπάρχει ωστόσο σημαντική βελτίωση της καταστάσεως και όπως είπα προηγουμένως μπορούμε να αποδώσουμε τη βελτίωση αυτή όντως στη βελτίωση των συστημάτων ελέγχου. Όσον αφορά την ανάκτηση ποσών που καταβλήθηκαν αδικαιολογήτως, υπενθυμίζω και πάλι ότι στην έκθεση αυτή τροποποιήσαμε την μεθοδολογία σε σύγκριση με παλαιότερα έτη και εναρμονίσαμε καλύτερα με τους εκδιδόμενου ετήσιους λογαριασμού. Δηλαδή τα ποσά που περιλαμβάνονται σε αυτή την έκθεση αναφέρονται στην εφαρμογή ε, δημοσιονομικών διορθώσεων καθώς και διαταγές ανάκτησης που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή. Τώρα, για να έχετε τη δυνατότητα να συγκρίνετε την κατάσταση με πέρσι, οι υπηρεσίε μου προέβησαν σε επανυπολογισμό των πληροφοριών το 2010 στη βάση της νέας μεθοδολογίας. Το δε αποτέλεσμα δείχνει ότι συνολικά η κατάσταση βελτιώνεται. Από 77% για τον αγροτικό τομέα έως 92% για δαπάνες που διαχειρίζεται ευθέως η Κομισιόν βελτιώνεται η ανάκτηση και 93% για την πολιτική συνοχής. Ε, οι δημοσιονομικές διορθώσεις που εφαρμόστηκαν είναι σημαντικές επίσης και υψηλότερες από το 2010. Ακόμα και αν υπάρχει μείωση του ποσοστού ανάκτησης για τον αγροτικό τομέα. Το υψηλότερο ποσοστό ανάκτησης ανεβρίσκεται στην πολιτική συνοχή και κυρίως λόγω του κλεισίματος της προγραμματικής περίοδου 2000-2006. Από την πλευρά των εσόδων, τα αποτελέσματα των, της, των ανακτήσεων των παραδοσιακών ιδιών πόρων μένουν περίπου σταθερά από χρόνο σε χρόνο και βελτιώνονται από 46% ε, το 2010 σε 52% το 2011. Συνολικά, 92% των χρεών των ιδίων πόρων που καθορίζονται κάθε χρόνο ανακτώνται χωρίς σημαντικά προβλήματα και σε εύλογο χρονικό διάστημα, δηλαδή μέσα σε περίοδο περίπου τριών ετών από τον καθορισμό του. Σε περιπτώσεις όπου τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, εκεί είναι κυρίως εκεί όπου υπάρχει υπόνοια απάτης. Και συχνά αυτό οφείλεται στη μακρά διάρκεια των ποινικών διαδικασιών που βέβαια καθυστερούν και τη διαδικασία ανάκτησης. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πολιτική και τα μέτρα τα οποία έλαβε, έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2011 για να εντείνει τον αγώνα κατά των απατών. Το 2011 η Κομισιόν ενέκρινε την τροποποιημένη πρότασή της για την μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Αγώνα κατά της απάτης και εσείς εγκρίνατε πρόσφατα τα ε, πορίσματα της ε, συζήτησης για την πρόταση αυτή. Τον Ιούνιο του 2011 πλέον η Κομισιόν ενέκρινε νέα στρατηγική κατά των απατών που τη λέμε στα αγγλικά CAFS και η οποία στοχεύει ιδιαίτερα στην αποκάλυψη των απατών στο επίπεδο των ε, ε, υπηρεσιών, από το επίπεδο δηλαδή των υπηρεσιών της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βελτιώσαμε επίσης την κοινοποίηση και την συνεργασία μεταξύ ποινικού δικαίου και ερευνών. Τον Ιούλιο καταθέσαμε και πρόταση οδηγίας για το ίδιο θέμα. Το 2011 η Κομισιόν επίσης ζήτησε να στοχευτεί περισσότερο η προσπάθεια στην διαφθορά και από το 2013 η Κομισιόν θα υποβάλει αναδιετία έκθεση για τον αγώνα κατά της διαφθοράς. Επίσης αργότερα το 2011 υποβάλαμε τρεις προτάσεις οδηγιών για τον εξυγχρονισμό των κανόνων των δημοσίων προμηθειών για την πρόληψη μη υγιών επιχειρηματικών πρακτικών. Επίσης η Κομισιόν ενέκρινε κοινοποίηση, ανακοίνωση μάλλον, για το μέλλον του ΦΠΑ σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι απάτες και στον τομέα αυτό. Η έκθεση του άρθρου 325, όπως κάθε χρόνο, διαλαμβάνει και μέτρα που λαμβάνουν οι χώρες μέλη στον αγώνα τους για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην φετινή έκθεση το συγκεκριμένο αυτό θέμα εξετάζει σε βάθος και στοχεύει ιδιαίτερα τους ελέγχους των χωρών μελών για την καταπολέμηση παρατυπιών και απατών στην πολιτική συνοχής, περιλαμβάνοντας πληροφορίες και για ανακρίσεις και έρευνες, στρατηγικά μέτρα και πολιτικές που έχουν ήδη αναλυφθεί. Και στο παράρτημα θα βρείτε τις απαντήσεις των χωρών μελών. Τέλος, η έκθεση του 2011 περιλαμβάνει και πληροφορίες για το πώς, ποια συνέχεια έδωσαν οι χώρες μέλη στις συστάσεις που τους έγιναν στην έκθεση του 2010. Και με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας λέγω ότι τα περισσότερα από τα θέματα τα οποία είχαμε περιλάβει στις συστάσεις του 2010 έχουν δει βελτίωση και ιδίω για την ανάκτηση αδικαιολογήτως καταπληθέντων ποσών για το IMS, για τον ρυθμό συμμόρφωσης στον αγροτικό τομέα και τις, στατηγικές, τις εθνικές που έχουν εγκριθεί για τους ε, τελωνιακούς δασμούς. Βεβαίως χρειάζεται περαιτέρω πρόοδο σε σχέση με μικρό αριθμό ε, χωρών μελών. Για παράδειγμα, η Γαλλία δεν έχει κοινοποιήσει καμία περίπτωση δόλιας παρατυπίας στον χώρο της πολιτικής συνοχής. Η Κομισιόν έχει αναλάβει διμερεί, πρωτοβουλίε διμερείς πρωτοβουλίες για να ε, συζητήσει τα θέματα αυτά. Άλλε χώρε έχουν λάβει προληπτικά ή προκατακτικά μέτρα για να ε, ρυθμίσουν για ε, τα, της περίοδου του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου. Αξιότιμα μέλη, νομίζω ότι μπορούμε συνολικά να πούμε ότι το 2011 επιτελέσαμε πρόοδο και από την πλευρά της Κομισιόν και από την πλευρά των χωρών μελών. Ωστόσο, δεν μπορούμε να, ε, να επαναβαθούμε στις δάφνες μας. Υπάρχει ένας αριθμός περιπτώσεων, διότι ορισμένε χώρε μέλη εξακολουθούν να ε, ε, κοινοποιούν πολύ χαμηλού αριθμού δολίων παρατυπιών. Δεύτερον, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα μέτρα πολιτικής τα οποία προτείνει η Κομισιόν υιοθετούνται και εφαρμόζονται όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και τέλος, οι αναλύσεις δείχνουν ότι χρειάζονται ακόμα προσπάθειες ώστε να διατηρηθεί η πρόοδος αυτή και να αντιμετωπιστούν τα πιθανά αντίστροφα αποτελέσματα, μάλλον αρνητικές επιπτώσεις της σοβούσας κρίσης. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και ευχαρίστω να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Äh, Ευχαριστώ κύριε Σεμέτα για την έκθεση και για την μεγάλη προσήλωση με την οποία το παρουσιάσατε. Ξεκινάμε τώρα τη συζήτηση στην Επιτροπή και θα ήθελα να ξέρω ποιος θέλει να ξεκινήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μας είπατε στην εισαγωγή σας ότι αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα και έχετε δίκιο. Είναι σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδίως σε αυτή την δυσχερή οικονομική και πολιτική συγκυρία είναι εξίσου δύσκολο για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, γι' αυτό και καλωσορίζω τον ε, Επίτροπο και τον ευχαριστώ για την ομιλία του σήμερα το πρωί. Πολλές φορές επικεντρωνόμαστε μόνο στα κακά νέα και θα ήθελα να ξεκινήσω αναφέροντας διάφορους αριθμούς τους οποίους ε, ανέφερε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είπατε δηλαδή ότι μειώθηκε η οι παρατυπίες μειώθηκαν κατά 35% και χαιρετίζω καταρχήν ε, στην αρχή των συζητήσεών μας αυτό το θέμα. Ε, ε, επίσης δεν αμφιβάλλω ότι το 2010 για το 2010 όλα αυτά τα αποτελέσματα θα αντικατασπριστούν στο τέλος του προγράμματος και ε, βλέπουμε ότι ε, υπάρχει μείωση στο 10, το 11 και όπως είπατε και εσείς υπάρχει μία μείωση των αριθμών. Παρ' όλα αυτά πρέπει να ε, καλωσορίσουμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και όσον αφορά την ανάκαμψη και την δυνατότητα επανακτήσεως των δαπανών ε, θέλω να χαιρετήσω τις προσπάθειες οι οποίες γίνονται. Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεχώρισε τις δόλιες ε, ε, παρατυπίες και τις αθελείς και ε, αυτό συνάδει με τις ε, προτάσεις του ελεκτικού συνεδρίου. Προσπαθούμε δηλαδή να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό και ήταν σαφής ο διαχωρισμός αυτό στην έκθεσή σας σήμερα. Επίσης ε, υπάρχουν σε διάφορα κράτη-μέλη διάφορα ποσοστά. Ε, δεν είναι δυνατόν να ξέρουμε πόσο, ποιο ποσοστό των παρατυπιών είναι δόλιες ή όχι. Ε, χρησιμοποιείται ορισμένες μεθόδους, ορισμένες χώρες ε, δηλώνουν υψηλό ή χαμηλό ποσοστό παρατυπιών και ε, πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε μεθόδους για να παραβάλουμε τους αριθμούς και να παρουσιάσουμε ένα σύστημα ε, το οποίο να είναι αυτό που επιτρέπει να συγκρίνουμε πλήρως τα στοιχεία. Θα ήθελα λοιπόν ε, αυτά να ε, είναι σαφή και προσπαθούμε να εφαρμόσουμε μέτρα κατά της ε, διαφθοράς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασίζεται στα στοιχεία που στέλνουν τα κράτη κατά τρόπον ώστε να ολοκληρώσει μία πλήρη εικόνα της κατάστασης και για την πληρωμή των προγραμμάτων. Ε, θέλω λοιπόν να ρωτήσω τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για να καταλύσει πλέον υπόλογα τα κράτη και για την ανακοίνωση των παρατυπιών και για την μη ε, ανακοίνωση των παρατυπιών που υπάρχουν. Τι μέτρα πρέπει ίσως να προωθηθούν που ισχύουν ήδη σε ορισμένα κράτη-μέλη και θα μπορούσαν να επεκταθούν και σε άλλες χρόνες. Επίσης, ε, εσείς είπατε ότι ε, έχετε ε, ήδη κάνει διάφορες επαφές με τα κράτη αποδίδουν οι προσπάθειές σας και σχετικά με το IMS τι πρόκειται να κάνετε για να εξασφαλίσετε την πλήρη εφαρμογή του IMS σε όλα τα κράτη-μέρη και σχετικά με ε, ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη θα ήθελα να μας πείτε τι γίνεται διότι βλέπουμε ότι 92% των ε, ανακτήσεων επιτυχάνονται. και μόνο ένα μικρό, μικρό ποσοστό της εκατό έχει προβλήματα. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι μπορεί να γίνει διότι ε, υπάρχουν διάφορα προγράμματα δράσης και επικοινωνίες οι οποίες εφαρμόζονται αντί να υπάρχει μία στεναρά δράση θα ήθελα λοιπόν να ξέρω πώς ε, όλα αυτά μπορούν να προωθηθούν και πώς μπορείτε να μας ενημερώσετε για το τι κάνετε. Ευχαριστώ κύριε Βόγκαν. Ο επόμενος ε, είναι η κυρία Ήκλασεν. Ε, ε, ε, ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν στατιστικές, η κυρία Γκρέσλε, δεν υπάρχουν στατιστικές οι οποίες μπορούν να αποδώσουν αν δεν ξέρουμε γιατί μιλάμε. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για τα στοιχεία και ανησυχώ γιατί βλέπουμε μία αύξηση πολλών ανακοινώσεων. Χαίρεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι βελτιώνεται το σύστημα τη της, της, των ανακοινώσεων μετά πέφτει το ποσοστό των ανακοινώσεων και χαίρεται γιατί αποδίδει το σύστημα της εποπτείας και ούτω καθεξής. Υπάρχουν όμως θέματα που είναι ανησυχητικά διότι υπάρχει μία άνηση ανακοίνωση των ε, περιπτώσεων μεταξύ κρατών μελών και τι σκοπεύει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι λέγεται στην έκθεση ότι για την έκθεση του έτους 2010 η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο ζήτησαν ε, γιατί δεν έχουν λάβει απαντήσεις, ε, γιατί υπάρχουν τόσο λίγες ε, ανακοινώσεις. Για το 11 αντιλαμβάνομαι ότι συνεχίζει το πρόβλημα αυτό με αυτά τα κράτη. Οπότε το ερώτημα είναι τι θα κάνουμε για να το επιλύσουμε, διότι ε, το ίδιο συνεχίζει να διαιωνίζεται και για την επόμενη περίοδο του IMF. Επίσης ε, σχετικά με τις recoveries, τις ανακτήσεις. Ε, έχουμε χώρες που πάντοτε είχαν προβλήματα, όπως η Ιταλία. Η Ιταλία λέγεται στην έκθεση ε, έχει 43% των ε, ε, ποσών που θα έπρεπε να επιστραφούν, δηλαδή σχεδόν το μισό. Και με ενδιαφέρει το θέμα των ανακτήσεων διότι θα ήθελα να ξέρω καταρχήν τι γίνεται και δεύτερον πώς μπορούμε να προχωρήσουμε διότι ποιες είναι οι επιπτώσεις οικονομικής σχετικά με τις ανακτήσεις, με τις recovery για την Ελλάδα, για την Ιταλία, για πολλά κράτη, διότι ε, αντιλαμβάνομαι ότι τα προβλήματα διαιωνίζονται. Σας παρακαλώ ε, <clears throat> απευθύνεται σε έναν ε, σε κάποιον κύριο δίπλα της κυρία Γκρέσλε. Ε, όλα αυτά τα στοιχεία βέβαια είναι κάτι που μπορείτε να μας δώσετε γραπτά, αλλά είναι στοιχεία που μας ε, είναι πολύ χρήσιμα. Εγώ είμαι από την ε, περιοχή Σβάμπεν στη Γερμανία και ε, συνήθως είμαστε φιδωλοί με τους επένους μας αλλά θέλω να σας επενέσω για αυτό που κάνατε εσείς και η Επίτροπος Ρέντινγκ για να προωθήσετε τις οδηγίες σχετικά με το ποινικό δίκαιο που ήταν ένα μέτρο πραγματικά απαραίτητο να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε την απάτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό σας συγχαίρω και η πολιτική ομάδα του ΕΛΚ θα στηρίξει πάρα πολύ στεναρά αυτή σας την προσπάθεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Γκρέστρο, ο κύριος Κυρλακάκης. Uh, uh, σας ευχαριστώ, Επίτροπε. Εγώ θα ήθελα καταρχήν να δηλώσω ότι πιστεύω πως η Κομισιόν έχει αναβαθμίσει την προσπάθειά της κατά της διαφθοράς και της απάτης. Ιδιαίτερα όσον αφορά τα ευρωπαϊκά οικονομικά ε, συμφέροντα. Πιστεύω ωστόσο πως σε αυτή τη φάση χώρο απέχουμε από την επίτευξη οποιου οποιασδήποτε σημαντικής πρόοδου και θα σας δώσω ένα σύντομο παράδειγμα. Ας πούμε η προσπάθεια για τα τελωνία που γίνεται είναι πολύ έντονη. Ωστόσο, αν δείτε τα στοιχεία της Transparency International, με βάση δημοσκοπήσεις όπου έχουν ρωτήσει τον κόσμο αν έχει δωροδοκίσει οποιαδήποτε συγκεκριμένη με κυβερνητική, κυβερνητικό οργανισμό ή θεσμό, θα δείτε 600.000 μικροφακελάκια στον τομέα των τελωνίων κάθε χρόνο στην Ένωση. Το επαναλαμβάνω, διότι δεν είναι εύκολο να το, να το χωνέψει κανείς. 600.000 κόσμος, νοικοκυριά, αναφέρουν ότι όλο και κάτι δίνουν στα τελωνία. Έχουν δωροδοκίσει κάποιον. Κατά τη δημοσκόπηση που έκανε η Transparency International στη διάρκεια 2010-2011. Ίσως αυτά να είναι λάθος, ίσως ο κόσμος να έχει τρελαθεί και να λέει ότι δωροδοκεί ενώ δεν δωροδοκεί. <laughs> Ίσως να μην συνειδητοποιούμε καν το τι συμβαίνει και σε ποιο βαθμό μπροστά στα μάτια μας. Εγώ πιστεύω πως είναι ισχύ το τρίτο, πιθανότατα. Και όταν βλέπω ότι κράτη-μέλη όπως η Γαλλία, ίσως και μικρότερα, όπως η Μάλτα, λένε πως δεν υπάρχει καμιά παρατυπία δόλια σε όλο το χειρισμό των ε, κοινοτικών ε, χρημάτων, αρχίζω να πιστεύω πως η ανθρώπινη φύση έχει αλλάξει και ότι για κάποιο μυστήριο λόγο έχουμε μεταλλαχθεί σε κάποια κράτη-μέλη. Η ανθρώπινη φύση έχει μεταλλαχθεί σε κάποια κράτη-μέλη. Ωστόσο, στην πράξη αυτό που συμβαίνει είναι πως υπάρχει προστασία που είναι σαν τείχος, αλλά είναι ένα τείχος μη επανδρομένο που προστατεύει την τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Και θα μιλήσω για την Όλαφ, η οποία το 2011, είδα 178 νέες υποθέσεις. Όλες, το 99% αυτών, ε, σύμφωνα με το Γενικό της Διευθυντή, προέρχονται από πληροφοριοδότες. Δεν υπάρχουν δηλαδή ε, ε, έρευνες ίδιες πρωτοβουλίες σε τομείς όπου γνωρίζουμε πως υπάρχει μεγάλη διαφθορά και χοντρή διαφθορά θα λέγαμε. Διερευνούν μικρές πραγματικές υποθέσεις διότι κανείς δεν τους μίλησε για τις μεγάλες ε, υποθέσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και άρα δεν κάνουν τίποτα. Από τη στιγμή λοιπόν που ισχύει ο κανόνας της σιωπή στον τομέα σας και και από τη στιγμή που πληρώνει κανείς όλους τους συμμετέχοντες, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα σε πειράξει. Αυτό είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα της πολιτικής μας κατά της απάτης. Και πάλι, αυτό το λέω παρότι συγχαίρω την Επιτροπή γιατί κάνει πολλές προσπάθειες. Η πραγματική ευθύνη για την, ε, για την καταστολή της απάτης είναι, ε, επιβαρύνει τα κρατημέλη, όπου δεν κάνουν τίποτα. Πιστεύω πως θα πρέπει να αναβαθμιστούν οι πολιτικές ε, κατά της διαφθοράς με, κατά τάξεις μεγέθους, αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή, γιατί στον νότο κόσμος μισεί αυτούς που κλέβει χρήματα από την Ένωση, γιατί τώρα αισθάνονται ότι τα κλέβουν από τους ίδιους. Ε, και στο Βορρά ο κόσμος δεν θέλει να πληρώσει πια στην Ένωση, γιατί πιστεύει πως ε, τα χρήματα αυτά δεν δαπανώνται σωστά. Πραγματικά λοιπόν πρέπει να επιταχύνουμε, τις, να αναβαθμίσουμε τις προσπάθειές μας, έτσι ώστε αυτοί που σκέφτονται να βουτήξουν χρήματα από την Ένωση να το ξανασκεφτούν πριν το κάνουν, γιατί αυτή τη στιγμή δεν το σκέφτονται ούτε καν μια φορά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σκυλακάκη. Η επόμενη ερώτηση του κυρίου Σμιτ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όλοι σε αυτό το κτίριο θέλουμε τα χρήματα μας να δαπανώνται με το σωστό τρόπο. Αυτό που εγώ θέλω να σας ρωτήσω αφορά τους πληροφοριοδότες, γιατί αυτοί είναι ε, πολύ σημαντικοί σε αυτούς τους τομείς που συζητάμε. Ο κύριος Κέσλερ λέει εδώ ότι υπήρξε μια μείωση των πληροφοριών που προέρχονται από δημόσιους ε, ε, από δημόσιες πηγές και έχει αυξηθεί η ενημέρωση από ιδιωτικούς φορείς και διερωτώ με γιατί. Άκουσα ότι όλοι φοβούνται για τη δουλειά τους και δεν τολμάνε να πούν τίποτα. Και αυτό ισχύει ε, όλος ιδιαίτερος για τα θεσμικά όργανα εδώ τη Ένωση. γιατί όπω ξέρετε είναι το χρυσό κλουβί, γιατί αν πεις κάτι, αν μαρτυρήσεις κάτι, θα αποκαλυφθούν όλα και σχετίζονται και με την δουλειά σου ε, άμεσα. Εγώ έχω διατελέσει το υπάλληλο στο δημόσιο τομέα και θα μπορούσα να επικρίνω το αφεντικό σα και να πω ότι δεν ισχύουν, δεν είναι όπως πρέπει τα πράγματα, αλλά εγώ θέλω να ακούσω τα σχόλιά γιατί είναι πολύ εύκολο να λέμε μειώθηκαν, αυξήθηκαν κτλ. Εγώ πιστεύω ότι αυτά όλα σχετίζονται με κάτι άλλο και όχι με... και με τα όσα είπε ο κύριο Κυλακάκη. Ευχαριστώ. Γκάιερ. Επόμενη ερώτηση, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, κύριε Σεμέτα, χαίρομαι για τα καλά νέα τα οποία μας έδωσε η έκθεση για τα, την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των κοινοτήτων εφέτος. Αλλά έχω τις ίδιες ανησυχίες όπως η συνάδελφος κρέσλε. Είμαι ε, ένας ε, ναυτικός, ιστιοπλώος και όταν είναι κανείς ε, σε ταραγμένες θάλασσες δεν είναι πάντοτε πολύ σκόπιμο να έχουμε τα πανιά όλα ανοιχτά διότι μπορεί να καταλήξει κανείς και να προσαράξει στη, στη ξηρά. Μπορούμε δηλαδή να προχωράμε πλησιστή και ε, να μην αντιληφθούμε ότι στο τέλος ε, δεν έχουμε προχωρήσει προς τη σωστή κατεύθυνση. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε κατά τη γνώμη σας, κατά τρόπον ώστε να έχουμε αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με το μέγεθος της απάτης διότι εμείς βασιζόμαστε στα κράτη-μέλη. Πολλοί συνάδελφοι μας είπαν ότι οι αριθμοί πότε είναι αξιόπιστοι και πότε λιγότερο. Το 0% απάτης με οδηγεί σε γιατί τότε ο κόσμος θα ήταν θαυμάσιος αν όλες οι χώρες μπορούσαν ε, να δηλώνουν ε, αξιόπιστα 0% αλλά εγώ ακολουθώ διαφορετική κατεύθυνση στη σκέψη μου ε, και γι' αυτό και πεθέτω την ερώτηση. Έχει κάποια πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μπορεί να μας πει τι πρέπει να γίνει κατά τρόπον ώστε να έχουμε αξιόπιστους αριθμούς σχετικά με την ε, κάλυψη της απάτης. Έχετε σκεφτεί τι μπορεί να γίνει με μελέτες της κοινωνίας των πολιτών σαν αυτές τις οποίες ε, πρότεινε ο κύριος Χιλακάκης. Έχετε κάποια πρόταση την οποία θα μπορούσαμε να απαιτήσουμε σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τα κράτη-μέλη κατά τρόπον ώστε πράγματι να έχουμε ένα σταθερό σημείο αναφοράς και να γνωρίζουμε ακριβώς εάν κινούμαστε ε, με το ιστιοπλοϊκό μας προς την ε, σωστή ε, κατεύθυνση για να πατάξουμε την απάτη ή θα προσαράξουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σοντή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Κύριε Γενική Διευθυντά, για αυτές τις εκθέσεις οι οποίες είναι πολύ σημαντικές. Καταρχήν σας ευχαριστώ διότι κατευθύνατε τις, τις εργασίες σας σε ένα διαχωρισμό μεταξύ της απάτης και των σφαλμάτων διότι άλλος είναι ο, ο αγώνας κατά της απάτης και άλλο κατά των σφαλμάτων διότι ξέρουμε ότι ουδής είναι αλάνθαστος και χαίρομαι που κάνατε αυτό το διαχωρισμό στην έκθεσή σας διότι ε, με εξέπληξαν οι σημαντικές ε, αυξομοιώσεις οι οποίες διαπιστώθηκαν σε αυτή την έκθεση όπου βλέπουμε ότι υπάρχει μία μείωση των ε, δηλώσεων για πάτες και ε, παρατυπίες και εφόσον ε, υπήρξε ε, μία έκθεση για το 2000-2006 όπου είδαμε τα αποτελέσματα των παρατυπιών το 2009 και 10 και εκεί βασίστηκε η έκθεση τώρα του 2011 Βλέπουμε λοιπόν μία μείωση ε, των ε, ανακοινώσεων παρατυπιών και δεν θα ήθελα ε, στα πλαίσια των εργασιών μας να σκεφτούμε ότι και να πιστέψουμε ότι υπάρχουν λιγότερες παρατυπίες στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ αυτό ίσως είναι απλώς μία αλλαγή προγραμμάτων αν δηλαδή το θέμα είναι ουσιαστικό ή απλώς ε, θέμα τυπικό παρουσίασης. Ε, υπάρχουν ε, τεχνικές, οι διορθωμένες στατιστικές των εποχικών αυξομοιώσεων, διακυμάνσεων για να μπορέσουμε να γνωρίζουμε μέσα ή στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ποια είναι τα επίπεδα της της απάτης. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι θα ήθελα να υπάρχει μία στατιστική για τις καταδίκες, άπαξ δηλαδή και ανακοινωθούν αυτές οι παρατυπίες και έχουμε στοιχεία ε, για τις, ε, τις επιστροφές πρέπει να γνωρίζουμε ε, πόσα πρόστιμα, πόσες καταδίκες για φυλάκιση, ποιοι είναι αυτοί που διέπραξαν τις παρατυπίες, αν είναι λογιστές, ελεγκτές, υπάλληλοι, ποιοι είναι δηλαδή δηλαδή τα στοιχεία και δεύτερον ποια ήταν η ποινική ε, συνέχεια σε αυτή τη διαδικασία αν υπήρξαν αθώσεις ή διαπιστώσεις όπου δεν υπήρχε ε, καμία ε, αξιόπινη πράξη. Και να ολοκληρώσω λέγοντας ότι θα ήθελα να αναρωτηθούμε σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σχετικά με την ε, κοινή διαχείριση διότι βλέπουμε ότι σε αυτή την έκθεση για τις παρατυπίες βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, μικρά ποσοστά όσον αφορά την μεμονωμένη διαχείριση και περισσότερα, πολύ περισσότερα σχετικά με την κοινή διαχείριση ως προς τα ποσοστά των παρατυπιών και αντιλαμβάνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα με τον οικονομικό έλεγχο και πρέπει να σταματήσουμε αυτή την κοινή διαχείριση διότι δηλαδή ήταν κάτι που ήταν χρήσιμο όταν είχαμε 5-6 κράτη, όταν δεν θέλαμε να έχουμε ε, μια ευρωπαϊκή ε, υπηρεσία δημοσίων υπαλλήλων, αλλά θα ήθελα να ξέρω τώρα ποιο είναι το κόστος, ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής ε, της κοινή διαχείρισης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και κρατών και μήπως δεν έφτασε η στιγμή να έχουμε τη δικιά μας διαχείριση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 την αρμόδια οικονομική διεύθυνση που ασχολείται με τις παρατυπίες διότι ε, το κερασάκι στην τούρτα είναι ότι οι Υπουργοί Οικονομικών δεν κατάφεραν να αυξήσουν ε, την, ε, και να βελτιώσουν τα οικονομικά των κρατών σε αυτή την κοινή διαχείριση και στα 8 δισεκατομμύρια τα οποία δεν ε, ε, μπόρεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανακτήσει τα ποσά αυτά και δεν μπορεί να πληρώσει τους λογαριασμούς τους οποίους χρωστάει και ε, οι υπουργοί είναι ανίκανοι και μετακυλούν τις ευθύνες από τη μια χρονιά στην άλλη και τώρα μιλούν για το 2012. Οπότε ε, πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση στο Κοινοβούλιο για την ε, γενική ε, οικονομική διαχείριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να σκεφτούμε από μια νέα οπτική γωνία να δούμε τι κοστίζει η κοινή αυτή διαχείριση και σας ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα έκθεση. Ο κύριος Μάουρο. Α, λάθος. Ο κύριος Μόλτερ. Ε, εξ είχαμε ένα από τους πιο σημαντικούς πόρους ε, του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον ε, ΦΠΑ και μπορεί να αποτελέσει και πάλι το ίδιο σημαντικό πόρο. Ξέρουμε πως η Κομισιόν εργάζεται για ένα μόνιμο φόρουμ για τις υπηρεσίες φορολόγησης, ώστε, ε, τις εφορίες, ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματικός ο ΦΠΑ. Γιατί όμως το κάνετε πολύ πιο γρήγορα, γιατί κατά τη γνώμη μου ο ΦΠΑ που είναι, είναι ένας εύκολος στόχος για πάτη και έπρεπε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα. Για ποιο λόγο ξεκινά αυτή τη στιγμή η Κομισιόν και μέχρι ποιο βαθμό θα προχωρήσει, ποιο σημείο θα προχωρήσει. Ευχαριστώ κύριε Μούλτερ και τώρα δίνω το λόγο στον Επίτροπο Σέμετα για να απαντήσει σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Φυσικά είναι μεγάλη ποικιλία των ερωτήσεων και σας ευχαριστώ. Να ξεκινήσω με τα γενικότερα στοιχεία. Ο κύριος Όντι με ρώτησε ποια είναι τα αίτια των ε, διακυμάνσεων. Προσπάθησα αυτό να το εξηγήσω στην αρχική μου ε, παρουσίαση γιατί με τη διαχείριση των κοινοτικών ταμείων έχουμε βεβαίως ένα κυκλικό φαινόμενο όπως το λέμε και γι' αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη συστήματα πολιετούς διαχείρισης και ελέγχου. Είναι φυσιολογικό λοιπόν ότι στο τέλος της δημοσιονομικής περίοδου, το τέλος της χρήσης, όταν τα προγράμματα βρίσκονται σε φάση κλεισίματος, όλοι, γίνονται τότε όλοι οι έλεγχοι. Αυτό έχει συμβεί το 2010 όταν ολοκληρώθηκαν τα προγράμματα 2000-2006 και αυτό βεβαίως ε, οδήγησε στην αύξηση των αναφερθησών παρατυπιών και απατών. Οπότε τώρα αυτή η προγραμματική περίοδος έχει τελειώσει και τα στοιχεία του 2011 δεν επηρεάστηκαν από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Εν μέρει λοιπόν έτσι εξηγείται η μείωση στο επίπεδο σφάλματος. Ένα άλλο μέρος οφείλεται στις βελτιώσεις του συστήματος ελέγχου και διαχείρισης, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα δράσης ε, για την πολιτική συνοχής ε, έχει εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια των περασμένων ετών και αυτό ε, έχει ε, φέρει αποτελέσματα όσον αφορά την καλύτερη κατάσταση στον τομέα των απατών. Τώρα, αν θέλουμε να δούμε συγκεκριμένα ζητήματα. Γιατί τέθησαν κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις σε σχέση με το τι πρέπει να κάνουμε ώστε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Εγώ πιστεύω πως είμαστε σε μια φάση όπου παρουσιάζονται πολύ σημαντικές ε, πρωτοβουλίες όπως αυτή της κυρίας Γκρέσλε για την προστασία των ευρωπαϊκών συμφερόντων μέσω του ποινικού δικαίου διότι πρέπει να κατανοήσουμε πως υπό την ισχύουσα νομοθεσία η Όλαφ έχει διοικητική λειτουργία, διοικητικού τύπου λειτουργία και οι ποινικέ κυρώσεις δεν είναι εναρμονισμένες, δεν έχουμε καν ε, καινούς ορισμούς για ποινικέ κυρώσεις και αυτό οδηγεί σε προβλήματα. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε σύντομα και ταχύτατα σε αυτούς τους τομείς. Μόλις έρχομαι από τη Γερμανία, το έχω συζητήσει με τις γερμανικές αρχές αυτό το θέμα, γιατί πιστεύω πως χωρίς τέτοιο είδους νομοθεσία φυσικά είναι πολύ πιο δύσκολο να προχωρήσουμε και να προχωρήσουμε κυρίως στην ποινική παρακολούθηση των ε, απατών. Έχουμε το μέσο όρο 42% νομίζω των υποθέσεων που υποβλήθηκαν από την Όλαφ στις Εθνικές Δικαστικές Αρχές, οι οποίες, ε, <clears throat> στις οποίες δόθηκε συνέχεια. Αυτό είναι μια παρατήρηση. Μια άλλη παρατήρηση είναι ότι αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε για μια νέα πρωτοβουλία για το μέλλον του Ευρωπαίου εισαγγελέα. Ε, έτσι θα δημιουργηθεί ένα ε, πολύ σημαντικό πολύ σημαντικό στοιχείο όσον αφορά την ποινική ε, δίωξη. Το αναφέραμε, για, προβλέπεται για τον Ιούνιο του 2013 και όσον αφορά τις νομοθετικές μας δράσεις νομίζω πως είμαστε στη σωστή πορεία αλλά θα πρέπει φυσικά αυτά να στηριχθούν και από αυτό το κοινοβούλιο ε, για να υιοθετηθεί ο κανονισμός περί Όλαφ, που πιστεύω πως έχει επίσης ε, σημαντικά βελτιωθεί. Και θα βελτιώσουμε τη σειρά την αποτελεσματικότητα της Όλαφ. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του εισηγητή, δηλαδή τι πρότυπα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, ποια μοντέλα που υπάρχουν στα κρατημέλη, Νομίζω πως αυτά τα θεματικά ερωτηματολόγια που στέλνουμε κάθε χρόνο φέτος αφορούσε τις δράσεις για την πολιτική συνοχής, το ερωτηματολόγιο αυτό δίνουν μια καλή ευκαιρία στα κρατημέλη να να δουν το ένα το άλλο και να μάθουν από τις καλές πρακτικές και να τις υιοθετήσουν. Πρόθεσή μας είναι λοιπόν να συνεχίσουμε αυτές τις πρακτικές με συγκεκριμένα θέματα, να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες για συγκεκριμένα ζητήματα. σε σχέση με τις ε, συνεδριάσεις που οργανώνουμε με τα κράτη-μέλη και μιλώντας γενικότερα Πιστεύω πως υπάρχει μεγάλη προστιθέμενη αξία σε αυτές τις επαφές, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να ε, δεσμευθούν και να κάνουν δραστηριότητες που σχετίζονται με την καταπολέμηση της απάτης. Εγώ πιέζω τις υπηρεσίες μου να... Ε, εργάζονται πιο εντατικά μόλις έρχονται πίσω από αυτές τις συνεδριάσεις να με ενημερώνουν διαρκώς για το εξελίξεις. Κράπια, κρατημέλη, Γαλλία και άλλοι που αναφέρουν σχετικά χαμηλά, χαμηλά νούμερα και στοιχεία. Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις σας ότι δηλαδή γι' αυτό το λόγο κιόλας οι υπηρεσίες μας δουλεύουν διμερώς με αυτά τα κρατημέλη και τώρα συνεχίζεται η συνεργασία με την Γαλλία. Ίσως ο Τζοβάνι Γκέσλερ θα μπορούσε να σας τα εξηγήσει πιο λεπτομερώς τι κάνουμε, αλλά αυτό το στοιχείο θα πρέπει να το δούμε από τη στιγμή που θα μπορούμε να καταλάβουμε κατά πόσο αυτά τα χαμηλά νούμερα που αναφέρουν κάποια κρατημέλη οφείλονται στον, όντως στον χαμηλό αριθμό απατών, στα θαύμα ή στην αποτελεσματικότητα των ε, αναφορών τους. Μέσα πάση περιπτώσει πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τα όρια για τα όσα μπορούμε να ζητήσουμε από τα κρατημέλη, γιατί έχουμε συγκεκριμένη νομοθεσία, αυτή μπορούμε να την, ε, ε, να την ακολουθήσουμε, μπορούμε να ζητήσουμε παραπάνω πληροφορίες, αλλά δεν μπορούμε να ζητήσουμε όποιες πληροφορίες θέλουμε. Μόνο αυτές που προβλέπονται από την νομοθεσία. then, regarding issues, issues Τώρα, σε σχέση με τη διαφορά και συγκεκριμένες έρευνες για την διαφθορά. Θα πρέπει να καταλάβουμε σαφώς ότι οι περισσότερες δράσεις εδώ πρέπει να γίνουν από τα κράτη-μέλη. Στο επίπεδο της Κομισιόν έχουμε γκρίνει ανακοινωθέν για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η διαφθορά πέρυσι. Για πρώτη φορά Έχουμε εισάγει επίσης τις ε, εκθέσεις από, την, ε, από τα κρατημέλη έτσι ώστε να υπάρχει πιο αντικειμενική ενημέρωση και να μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις και σύγκριση επιδόσεων των κρατών μελών. Πιστεύουμε πως αυτό θα οθήσει τα κρατημέλη σε βελτιώσεις στα συστήματά τους, στις νομοθεσίες τους. Γιατί κανείς δεν θέλει να βρίσκεται πάνω-πάνω σε αυτή τη θέση για το συγκεκριμένο θέμα. Σε σχέση με τις έρευνες της Όλαφ και το γεγονός ότι οι περισσότερες ε, οφείλονται σε εκθέσεις πληροφοριοδοτών ή ε, ε, άλλες πηγές. Συμφωνώ ότι αυτό είναι πρόβλημα. Και πιστεύω ότι με την έγκριση της μεταρρύθμισης της Όλαφ, δηλαδή αφού μεταρρυθμιστεί η σχετική νομοθεσία, θα στραφούμε σε περισσότερες δράσεις ίδιας πρωτοβουλίας. Και εγώ αυτό θα επιθυμούσα, γιατί τώρα... Μόνο μετά από αναφορά οφείλουμε να αντιδράσουμε. Πάντως πιστεύω πως μια καλύτερη χρήση της πληροφορίας, ε, καλύτερη ενημέρωση θα πρέπει να είναι η προτεραιότητα για τις μελλοντικές δραστηριότητες της Όλαφ. Τώρα, σε σχέση με το θέμα των πληροφοριοδοτών, Φυσικά δεν είναι εύκολο να εξηγήσουμε γιατί έχει συμβεί, αλλά θα πρέπει να σας πω ότι η Κομισιόν θα υποβάλει πρωτοβουλία σε σχέση με τον τους πληροφοριδότες. Σκοπεύουμε να υιοθετήσουμε και μια εσωτερική στρατηγική επί του θέματος αυτού μέχρι τα τέλη του έτους. Νομίζω ότι πρέπει να δημιουργήσουμε όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να εξασφαλίσουμε πως οι πληροφοριδότες προστατεύονται πλήρως από οποιαδήποτε δράση εναντίον τους. Νομίζω πως ε, αυτό θα βρίσκεται και στην καρδιά της μελλοντικής μας πολιτικής. Τώρα, για την ερώτηση του κ. Οντή για την κοινή διαχείριση και την ιδέα του ε, να μετατραπεί αυτή σε άμεση διαχείριση. Ξέρετε ότι αν λάβουμε υπόψη τους περιορισμένους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας, ε, καθώς και τις δεσμεύσεις της Κομισιόν και άλλων θεσμικών οργάνων να μειώσουν τον αριθμό του προσωπικού τους με το 2017, αν θυμάμαι σε μεγάλο μάλιστα βαθμό, νομίζω πως είναι αδύνατον να υλοποιηθεί, διότι υπάρχει πολλοί κόσμος στο κράτη-μέλη που ασχολείται με τη διαχείριση και τον έλεγχο των, κοινών, των ταμείων Κοινής διαχείρισης και Γι' αυτό θα πρέπει να επιμείνουμε στις βελτιώσεις, στην κοινή διαχείριση. Και μπορώ να επαναλάβω άλλη μια φορά αυτά που είπα όταν ε, σας ε, παρουσίασα την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό δηλαδή σε μια νομοθεσία ιδιαίτερα στην νομοθεσία περί των ε, ταμείων συνοχής, περί του Ταμείου Συνοχής ότι είναι πολύ σημαντικό οι προτάσεις που παρουσιάζονται με βάση αυτή την νομοθεσία όσον αφορά την, ε, τους όρους, ε, όσον αφορά τους ελέγχους να παραμείνουν όλα αυτά μέσα στην νομοθεσία γιατί αυτό θα βελτιώσει την κοινή διαχείριση, την μεικτή διαχείριση σε σχέση με την ισχύουσα κατάσταση. Οι αλλαγές σε αυτό το τομέα είναι δύσκολο να προβλεφθούν. Σε σχέση με την στατιστική και το ε, φάσμα το οποίο καλύπτει. Εμείς συλλέγουμε τις στατιστικές που προβλέπονται από την νομοθεσία και αυτό είναι η ουσία της έκθεσής μας, αλλά σας διαβεβαιώ και συμφωνώ μαζί σας ότι θα είναι ενδιαφέρον να δούμε ε, τα τελικά αποτελέσματα αυτών των ε, ερευνών θα μπορούσαμε να συζητήσουμε με τα κράτη-μέλη αν είναι δυνατόν να έχουμε τις πληροφορίες από εκείνα, αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο επί θελούσιας βάσης γιατί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπεται η παροχή τέτοιων πληροφοριών. Σε σχέση τώρα με το σύστημα διαχείρισης των παρατυπιών, Το θέμα είναι πόσο καλά χρησιμοποιείται. Η ερώτηση μάλλον ήταν αυτή. Θα πρέπει να σας πω ότι... Ε, χρησιμοποιούνται με αποτελεσματικό τρόπο, αλλά υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που δεν χρησιμοποιούν πλήρως τα πλεονεκτήματα του συστήματος διαχείρισης παρατεπιών. Και αυτό το ξέρω λόγω των διμερών επαφών που σας ανέφερα όπου προσπαθήσαμε να επιστήσουμε την προσοχή των κρατών μελών σε αυτό το εργαλείο που υπάρχει ήδη και του ζητήσαμε να το χρησιμοποιούν με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Ελπίζω λοιπόν έτσι να κάλυψα όλες τις ερωτήσεις που προέκυψαν κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης. Και φυσικά, φυσικά όταν ε, τα στοιχεία είναι καλύτερα, όπως είπε και η κυρία Γκρέσλε, υπάρχουν πάντοτε ερωτήματα το γιατί βελτιώνονται και όταν ε, τα πράγματα πάνε χειρότερα ε, τα ρίχνουμε όλα στο, το φταίξιμο στην Κομισιόν. Φέτος έχουμε καλύτερη κατάσταση και το, αυτό που μπορώ να επαναλάβω είναι ότι φυσικά υπάρχει κυκλικό, υπάρχουν μάλλον κυκλικά φαινόμενα τα οποία επηρεάζουν αλλά είναι εξίσου σημαντικό να δούμε την επιρροή του Κοινοβουλίου και αν δούμε κάπως ευρύτερα τις προοπτικές πέρα από το PDP, θα δούμε ότι υπό το ισχύον PDP είμαστε χαμηλότερα σε όγκο παρατυπιών από ό,τι παλιότερα, άρα προχωράμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Όντως θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα, αλλά Είναι πολύ σημαντικό για το λόγο αυτό το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να υιοθετήσουν τις προτάσεις που υποβάλαμε και τώρα έχουμε πολύ σημαντικές προτάσεις επιτάπητος. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπη που θέσατε υπόψη μας τις απόψεις σας για αυτό το σημαντικό θέμα, πώς δηλαδή να βελτιωθεί η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ενώσεως. Τώρα, ο εισηγητής επιθυμεί να λάβει το λόγο για την ολοκλήρωση γιατι αλλιω αλλιώς επειδή έχουμε περίπου 15-20 λεπτά να δώσω το λόγο στον κύριο Κέσλερ και να... Ναι, λίγα λόγια ως συμπέρασμα, ας πούμε, στην ε, παρουσίαση του Επιτρόπου. Οι συνάδελφοί μου έθεσαν σημαντικές ερωτήσεις και νομίζω ότι καλώς απήντησε ο Επίτροπος και λεπτομερός. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα και που είπαν και άλλοι, ότι δηλαδή θα πρέπει να μας ικανοποιεί η βελτίωση των αποτελεσμάτων αλλά οι συνάδελφοί μου θέλουν να γνωρίζουν και τους λόγους για τη βελτίωση αυτή. Δεν αμφισβητούμε τους αριθμούς που μας δώσατε. Θέλουμε να γνωρίζουμε ποιες είναι οι αιτίες που προκάλεσαν την βελτίωση αυτή, ώστε να συνεχίσουμε την ίδια προσπάθεια στο μέλλον. Επίσης, η διαφορά στους μηχανισμούς κοινοποίησης των παρατυπιών ανάμεσα στις χώρες μέλη που οδηγεί και σε διαφορά αποτελεσμάτων, σε διαφορά δηλαδή αριθμών περιπτώσεων. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί το δυνατόν ταχύτερο. Είναι ένα από τα θέματα που σημειώνω από τη σημερινή συζήτηση. Και γενικώ οι συνάδελφοί μου ενδιαφέρονται να γνωρίζουν πώς μπορούμε να ανακόψουμε την απάτη και στα έσοδα και στις δαπάνες. Και αυτά θα αποτελέσουν την βάση για τις συζητήσεις μας και στο μέλλον, που ασφαλώς θα συνεχίσουν να γίνονται Ευχαριστώ τους αδέρφους μου για τις, ε, για τις ερωτήσεις που σας έθεσαν και ευχαριστώ και εσάς για τις απαντήσεις που δώσατε. Ευχαριστώ κύριε Βόν, ευχαριστώ και τον κύριο Επίτροπο. Κύριε Κέσλερ, εσείς τώρα να ε, μας ε, κάνετε την παρουσίαση για την Όλαφ. Φαίνεται πως δεν έχουμε πολύ χρόνο. Λίγες λοιπόν σύντομε παρατηρήσει και είμαι στη διάθεσή σα αν θέλετε να μου θέσετε ερωτήσει. Και πρώτα είδατε την έκθεση. Ελπίζω ότι θα σας άρεσαν τα νέα γραφήματα. Κάναμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να γίνει πιο ευανάγνωστη η έκθεση, πιο ενημερωτική και πιο διαφανιστική. Και έτσι θα συνεχίσουμε κιόλας. Πέρσι ήταν μεταβατικό έτος για την Όλαφ. Από πέρσι αρχίσαμε την εσωτερική επανεξέταση της οργάνωσής μας που οδήγησε και σε αναδιοργάνωση και σε νέα ερευνητική διαδικασία που άρχισε να ισχύει από την 1η Φεβρουαρίου 2012. Παρ' αυτά, επιτρέψτε μου να τονίσω ορισμένα ενδιαφέροντα δεδομένα ε, που ε, συναποτελούν και κάποιες τάσεις που ίσως μπορούν να οδηγήσουν και σε κάποια συμπεράσματα ή πάντως κάποια συζήτηση και αποφάσεις. Όπως βλέπετε πρώτα, το 2011 η Όλαφ έλαβε συνολικά πάνω από χίλιες πληροφορίες που ενδεχομένω είχαν ενδιαφέρον για να ξεκινήσει μια έρευνα. Αυτό είναι ιστορικό ρεκόρ για την Όλαφ και δείχνει μια σταθερή τάση μέσα από τα χρόνια διότι η Όλαφ λαμβάνει όλο και περισσότερες πληροφορίες που ενδεχομένως έχουν ενδιαφέρον. Έχοντας φτάσει λοιπόν στο ιστορικό ρεκόρ το 2011 της 12 ετίας, φέτος, θα το ξέρουμε βέβαια του χρόνου ακριβώς στην επόμενη έκθεση, αλλά ήδη προβλέπω ότι φέτος, το 2012 δηλαδή, θα σπάσουμε το ρεκόρ αυτό και πάνω από 30%. Άρα, το 2012 κατά πάσα πιθανότητα θα φτάσουμε περίπου τις 1300 καταγγελίες. Αυτά τα νούμερα κάτι λένε και για την αντίληψη που έχει το κοινό για την Όλαφ, την ε, εμπιστοσύνη που δείχνει το κοινό και η εταίροι μας στην Όλαφ και βεβαίως αυξάνονται έτσι οι αιτήσει για διεξαγωγή ερευνών από την Όλαφ και είναι και ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά την αύξηση του ερευνητικού έργου της όλα. Ορισμένοι ήδη από εσά τονίσατε ότι υπάρχει και μια άλλη ενδιαφέρουσα τάση την οποία θα παρατηρήσουμε πολύ προσεκτικά και θα βάλουμε πιο λεπτομερείς στατιστικές τάση δηλαδή αύξησης των πληροφοριών προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα που περιλαμβάνει και επιχειρηματίες, εταιρείες, μεμονωμένους πολίτες και ανώνυμες πηγές και μία σταθερή μείωση εισερχόμενων πληροφοριών από αυτά που αποκαλούμε εμείς δημόσιες πηγές, δηλαδή αρχές των χωρών μελών και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα καθ' αυτά. Δεν μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι η τάση αυτή συνεχίζεται το 2012, αλλά από μια άποψη αυτή η τάση μας ενθαρρύνει, διότι δείχνει ότι γίνεται πιο γνωστή η Όλαφ στο κοινό, στους πολίτες, ότι έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη και επομένως και περισσότερη ανάγκη ενδεχομένω από την Όλαφ. Από την άλλη μεριά πρέπει να αναλύσουμε και αναχώρα μέλο, αναθεσμό, ε, τι γίνεται, τα έχουμε αρχίσει να τα κάνουμε αυτά. Να δούμε δηλαδή και ποιοι είναι οι λόγοι της μείωση της κοινοποίηση πληροφοριών από δημόσια όργανα. Δεύτερο, από όλες αυτές τις εισερχόμενες πληροφορίες, κάθε εισερχόμενη πληροφορία σημαίνει και το άνοιγμα ενός φακέλου. Έχουμε λοιπόν και έναν άλλο σταθερό αριθμό που θα δείτε και στην περσινή έκθεση. Άνοιξε 180 έρευνες η Όλαφ και αφού εργαζόμαστε στη βάση της αρχής της επικουρικότητας, προβαίνουμε σε επιλογή υποθέσεων. Δεν ανοίγουμε, δεν ξεκινούμε έρευνα για κάθε υπόθεση, ούτε άλλωστε κάθε πληροφορία, κάθε εισερχόμενη πληροφορία είναι ε, ουσιαστική και έχει κάποια θεμελίωση. Κάθε χρόνο λοιπόν η Όλαφ ανοίγει ένα αυξανόμενο αριθμό υποθέσεων και για το 2012 φαίνεται να πηγαίνουμε για ρεκόρ πάλι ανοίγματο φακέλων. Ήδη το 2012 από την 1η Φεβρουαρίου έχουμε ανοίξει 260 έρευνες μέχρι τέλη Οκτωβρίου φέτος. Και πάλι εδώ λοιπόν η Όλαφ τελειο οκτωβριου φετος και παλι εδω μέχρι το όριο, μέχρι το από το όριο της ικανότητάς της, ίσως να το ξεπερνά κιόλας. Για την αντιμετώπιση όχι μόνο όλων των εισερχόμενων πληροφοριών, αλλά και των συνεχιζόμενων ερευνών. Όπως είδατε στην περσινή έκθεση, είχαμε και άλλο ρεκόρ. Δεν έχουμε σταθερή τάση εκεί, σε ό,τι αφορά δηλαδή την δημοσιονομική ανάκτηση. Πέρσι υπήρξε ρεκόρ για διάφορους λόγους. Πρώτο διότι ήταν μεγαλύτερη η ανάκτηση που σήμανε αύξηση των εκατομμυρίων, των ανακτώμενων εκατομμυρίων, αλλά και αναφέρεται άλλωστε στην Ιταλία, αυτό το λέει καθαρά η έκθεση, αλλά και χωρίς αυτή την περίπτωση της Ιταλίας θα ήταν πάλι ρεκόρ ανακτήσεων η ανάκτηση. Τα εκατομμύρια, τα κονδύλια τέλο πάντων, καταγράφονται στις στατιστικές του έτους όπου γίνεται η ανάκτηση. Αναφέρονται όμως βέβαια σε έρευνα που έχει διεξαχθεί στο παρελθόν. Πάντως αυτό που μετρά είναι το σημαντικό οικονομικό όφελος και ότι τα σχετικά αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί από την Όλαφ σε απόλυτους δε αριθμούς ξεπερνούν το διοικητικό κόστος της Όλαφ. Το ξεπερνούν πολύ σημαντικό, σημαντικά. Είναι πολύ σημαντικά τα ποσά αυτά. Το ίδιο σημαντικό στοιχείο στην έκθεση, στο οποίο εφιστώ την προσοχή σας, πάλι ένα ρεκόρ σε ό,τι αφορά τις καταδίκες από τα δικαστήρια των χωρών μελών εάν δηλαδή το βάλουμε σε βάση ετών φυλάκισης που επέβαλαν οι εθνικές δικαστικές αρχές μετά από τα πορίσματα των ερευνών της Όλαφ. Ίσως τα νούμερα αυτά να μην είναι τόσο ελκυστικά, ούτε ευχάριστα, αλλά τέλος πάντων στο τέλος της υπόθεσης, όταν αποκαλύπτεται μια απάτη, χρειάζεται βεβαίως και την πρέπουσα αντίδραση από τις χώρες μέλη. Έτσι λοιπόν πέρσι είχαμε άλλο ένα ρεκόρ σχετικά. Εν τέλει, δύο σημεία, δύο θέματα ακόμη, για την πλευρά της πολιτικής. Η Όλαφ είναι γνωστή για την ερευνητική της ικανότητα, αλλά και από την πλευρά της πολιτικής, πώληση δηλαδή. Εδώ δεν μπορούμε να μετρήσουμε στη βάση των στατιστικών, αλλά σε ό,τι αφορά τον αριθμό πρωτοβουλειών πολιτικής και νομοθετικών πρωτοβουλειών, στις οποίες συμμετέχει ευθέως η ε, όλα, και αν δεν ηγείται πάντοτε των πρωτοβουλειών αυτών. Ωστόσο, τα δύο αυτά χρόνια φτάσαμε σε άλλο ιστορικό ρεκόρ. Οι άνθρωποι μας, των διευθύνσεων πολιτικής, βεβαίως και με συνεργασία με άλλα θεσμικά όργανα, και σε ό,τι αφορά την επεξεργασία της προαναφερθήσης οδηγίας για το ουσιώδες ποινικό δίκαιο, για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπου οι σχετικές προτάσεις εγκρίθηκαν τον Ιούλιο από την Κομισιόν, αλλά βέβαια συνεχίζουμε την εργασία μας και απέναντι στα άλλα θεσμικά όργανα. Η Όλαφ επίσης εργάζεται για την επεξεργασία νέας νομοθεσίας για παραχάραξη νομισμάτων ευρώ, καθώς και για την αναθεώρηση του κανονισμού 515 για την αμοιβαία αρρωγή στον τομέα των τελωνίων. Και έχουμε συμμετάσχει και, στην, και στο σχεδιασμό της πρότασης για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καπνών και προϊόντων, καπνού και προϊόντων καπνού στα ανατολικά σύνορα. Και Συνεργαζόμαστε επίση στην εκπόνηση του εγγράφου της Κομισιόν για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προϊόντων καπνού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια ένα πολύ σημαντικό θέμα αλλά και μεγάλη πρόκληση και πολλή δουλειά μαζί με την Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης για την πρόταση ΕΠΟ. Ε, επομένως, έχουμε δουλεύουμε και σε θέματα πολιτικής, πώληση δηλαδή, πάλι με τρόπο πρωτοφανή στην ιστορία της ε, Όλαφ. Άρα το προσωπικό μας και αυτό που ασχολείται με τις έρευνες, αλλά και αυτό που ασχολείται με την διαμόρφωση πολιτικής, δουλεύει όπως δεν έχει ξαναδουλεύει ποτέ στο παρελθόν. Και μέχρι το όριο των ικανοτήτων του, των δυνατοτήτων του καλύτερα. Τελειώνω σημειώνοντας ότι όλα αυτά βέβαια μέσα σε ένα πλαίσιο περικοπής ή περικοπών προσωπικού, διότι η Όλαφ έχει και το αρνητικό ρεκόρ των περικοπών του προσωπικού της, που δεν έχει ξανασυμβεί στην ιστορία της. Ήδη από φέτος όπως και σε όλες τις υπηρεσίες, σχεδόν σε όλες τις υπηρεσίες της Κομισιόν, μας επιβάλλονται περικοπές 2% ανά έτος για 4 χρόνια. Θα έχουμε λίγο λοιπόν πάνω λιγότερο προσωπικό και για τις δύο δραστηριότητες μας και έρευνα, οι έρευνες μάλλον και διαμόρφωση πολιτικής. Πάντως νομίζω ότι καλά τα έχουμε καταφέρει παρόλα αυτά μέχρι τώρα και θα συνεχίσουμε. Κάνουμε κάθε τι που μπορούμε για να ανταποκριθούμε άλλωστε και στην αυξανόμενη εμπιστοσύνη του κοινού απέναντι στην Όλαφ. Και όπως είπα και πριν, τα νούμερα που σας προανέφερα δηλαδή, το αποδεικνύουν. Ευχαριστώ κύριε Κέσλερ για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Στην ουσία έχουμε εξαντλήσει το χρόνο μας για το θέμα αυτό. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να ρωτήσω αν συνάδελφοί μου έχουν σχόλια ή ερωτήσεις και σύντομα να τις υποβάλουν στον ε, κύριο Κέσλερ, ο εισηγητής και η κυρία Γκρέσλερ. Κύριε Βόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λόγω του χρόνου, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον Γενικό Διευθυντή της Όλαφ για την ομιλία του και για την έκθεση. Γιατί δεν είναι πάντοτε εύκολο να καταστήσει κανείς ενδιαφέρον ένα τέτοιο θέμα και ευανάγνωστο. Αλλά νομίζω πως εδώ τα κατάφερε. Η έκθεσή του είναι πολύ ε, κατανοητή. Πρέπει να Είπαμε ήδη σήμερα το πρωί ότι προσπαθούμε όντως να περιορίσουμε τις ε, πάτες. Είναι σημαντικό θέμα για την Επιτροπή μας και ο Γενικός Διευθυντής έδωσε το παράδειγμα όσον αφορά την, το λαθρεμπόριο καπνού και ε, τσιγάρων. 90% των χρημάτων όταν ε, κατάσχονται τσιγάρα δεν πηγαίνουν ε, στα ίδια τα κρατη Και επίσης θα πρέπει να εστιάσουμε στην την προσοχή στην πολιτική συνοχή. Σίγουρα μιλάμε για αυτήν πολύ όταν παίρνουμε την ετήσια έκθεση του ε, ελεγκτικού συνεδρίου και εκεί είναι το θέμα της ε, πολιτικής συνοχής και της συνέπειας όσον αφορά την πολιτική μας για τις κρατικές προμήθειες, κρατικές συμβάσεις. Ε, θα είμαι λοιπόν σύντομος. Έχω να κάνω κάποιες ερωτήσεις ε, για τον Γενικό Διευθυντή. Η πρώτη είναι μια γενικού περιεχομένου ερώτηση. Ανέφερε ε, ότι είναι σημαντικό να δοθούν προτεραιότητες στις εργασίες της Όλαφ. Ε, σε ποια μέτρα λοιπόν πιστεύει ότι θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή στην προσπάθεια μείωσης των απατών. Αν έπρεπε να διαλέξει δύο-τρία πράγματα, ποια θα ήταν αυτά όσον αφορά τον μεγαλύτερο αντίκτυπο για την μείωση της απάτησης στην Ένωση. Επίσης, ε, Είπαμε ότι 75% των νέων περιπτώσεων προέρχονται από ιδιώτες, αλλά μόνο το 5 10% δηλαδή από αυτές ερευνάται. Ποιους μηχανισμούς χρησιμοποιεί λοιπόν η Όλαφ για να αποφασίσει ποιες από τις αναφορές είναι γνήσεις και ποιες θα διερευνήσεις. Ε, το τρίτο μου ερώτημα αφορά το τσιγάρα και το καπνό και το λαθρεμπόριο αυτό το οποίο ανέφερε ο Γενικό Διευθυντή και εγώ ανέφερα περιορισμένο, λέγοντα ότι είναι σημαντικό για το κρατη και για την Ένωση. Το ερώτημά μου είναι, έχει καθόλου βελτιωθεί η κατάσταση όσον αφορά το λαθρεμπόριο αυτών των προϊόντων. Για παράδειγμα, ε, μέσω εξάντε και εξπόστο ελέγχων και έπειτα, ποιε είναι οι πιθανότητε συνεργασία ανάμεσα στο όσα κάνει όλο αυτό το πρόγραμμα Hercule 3, Ηρακλή 3 και τα υπόλοιπα όλα προγράμματα θέματα, ποιες προσπάθειες συντονισμού γίνονται ώστε να έχουμε μεγαλύτερο αντίκτυπο στη μείωση του λαθρεμπορίου τσιγάρων και καπνού. Και τελευταία μου παρατήρηση είναι γενική φύση και αφορά τις, ε, άτυπες, ε, τις, ε, τις προτάσεις της Όλαφ. Τις ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής, αλλά έχω την εντύπωση ότι οι προτάσεις αυτές δεν είναι ιδιαίτερα ε, έγκυρες, ας πούμε το τεκμήριο αθότητας έπρεπε ήδη να υπάρχει εδώ. Επίσης η ανάθεση εντολή στην Όλαφ για να δουλέ, συνεργαστεί με άλλα ευρωπαϊκά σώματα και θεσμούς και συνεργασία με τρίτες χώρες, αυτά είναι θέματα κοινή λογικής. Ε, και γι' αυτό και η ερώτησή μου πάει στο Γενικό Διευθυντή θεωρεί ότι αυτές οι προτάσεις περί μεταρρύθμισης είναι αρκετές για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του στην Όλαφ. Η κυρία Γκρέσλο και ο κύριος Σκυλακάκης και τέρμα μετά. Ευχαριστώ. Τρεις ερωτήσεις προς τον Γενικό Διευθυντή. Καταρχήν ε, χαίρομαι διότι τουλάχιστον ε, ε, είναι ουσιαστική η έκθεσή του δυόμιση χρόνια θέτεται σαν μέσα μέσο όρο για κάθε ε, έρευνα ενώ αναφέρεται άλλος αριθμός ε, και έτσι θα ήθελα να ξέρω ε, γιατί αυξήθηκε κατά δύο μήνες ο χρόνος της έρευνας από το 2010 ως το 2011. Αυτό τουλάχιστον βλέπουμε στην έκθεση. Ε, ανατάχθηκε η υπηρεσία της Όλαφ και από τις έρευνες ε, διαβλέπουμε ότι στους τομείς που γίνονται ε, έρευνες υπάρχουν μονάδες με άτομα που δεν έχουν πείρα σε έρευνες πώς είναι δυνατόν δηλαδή να χρησιμοποιεί κανείς ε, ε, τέτοια άτομα υπάρχουν και νομικές παρατυπίες ή παραβάσεις νομικές πώς τις αντιμετωπίζει η Όλαφ μετά σχετικά με τα προϊόντα καπνού. Βλέπουμε και στην περίπτωση Νταλή ότι υπάρχει στενή σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της βιομηχανίας καπνού. Δεν απαγορεύεται αυτό, αλλά όταν υπάρχουν δύο ε, παρόμοιοι λογότυποι ο ένας δίπλα στον άλλον, ε, εμφανίζεται σαν να υπάρχει ε, κάποια χορηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τη βιομηχανία καπνού. Κύριος Χιλακάκης. Θα είμαι πολύ σύντομο. Ο Επίτροπος Σεμέτα είπε προηγουμένως ότι στις έρευνες ίδιες πρωτοβουλίες Ε, δεν, έχει, δεν, μπορεί να το κάνει ακόμα η Όλαφ. Ε, αναμένω λοιπόν πρόταση για το πώς πιστεύει ότι θα μπορέσει να το κάνει αυτό η Όλαφ, να πάρει τις ίδιες πρωτοβουλίες. Ε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν από κάποιε εβδομάδε, όταν ε, το Ελληνικό Συνέδριο υπέβαλε την έκθεσή του, μίλησε για 3,90% ποσοστό σφάλματο. Και εγώ ρώτησα τον κύριο Σεμέτα αν ε, αν θεωρούσε λογικό το αυξανόμενο αυτό ποσοστό. Και επανήλθε και μας είπε ότι υπήρχε ανάκτηση 1,2 το οποίο θα πρέπει να αφαιρέσουμε από το ποσοστό σφάλματος 3,9% και ότι δεν έπρεπε έτσι να το βλέπουμε. Με πάση περιπτώσει, εσείς είπατε ότι το σύνολο ανάκτησης είναι 19.600.000 ευρώ. Γιατί, σε πόσα χρόνια, για πόσα χρόνια μιλάμε. Γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε και να γνωρίζουμε το ποσοστό ετήσιας ανάκτησης. Σας ευχαριστώ. Μπορείτε να σχολιάσετε κύριε Κέσλερ για, σε μερικά λεπτά. Ναι, θα προσπαθήσω. Ο κύριος Βόν με ρώτησε ποιος μεχανισμός, αν και πώς θα αρχι... Ε, ε, ιεραρχήσουμε Βασικά ήταν περίπου το 1 πέμπτο της ενημέρωσης πάντα, της πληροφόρησης πάντα. Ναι, και δεν αναφέρεται στην έκθεση, διότι πρέπει να πω πως η έκθεση αναφέρεται στο 2011. Εγώ ανέλαβα τα καθήκοντά μου στη διάρκεια του 2011 και ξεκινήσαμε εσωτερική αναθεώρηση, η οποία οδήγησε σε μεγάλες αλλαγές που έγιναν μέχρι την πρώτη ε, Φεβρουαρίου 2012. Από αυτές τις αλλαγές μια από τις πιο σημαντικές ήταν ακριβώς το θέμα της διαδικασίας επιλογής και ιεράρχησης για την έναρξη ή μη μιας ε, έρευνας. Το 2011 όλα αυτά είχαν αφαιθεί στην ερευνητική μονάδα, δηλαδή δεν υπήρχε κάποιο μέσο κάποιο, για, να, διαχειριστούμε την έναρξη της έρευνας με συνεπή τρόπο. Ε, από την 1η Πρώτου 2012 έχουμε μια ειδικευμένη μονάδα, την μονάδα επιλογής που λαμβάνει με διαφανή τρόπο όλες τις εισερχόμενες πληροφορίες ενδεχόμενου ερευνητικού ενδιαφέροντος και δίνει στον Γενικό Διευθυντή τη γνωμοδότησή της αφού έχει προβεί σε κάποια επιλογή για την έναρξη μη κάποιες ίδιες έρευνας ή έρευνα ίδιες πρωτοβουλίες ή με βάση κριτήρια τα οποία είναι δημοσιευμένα και άρα διαφανή υπάρχουν στο website μας. Φυσικά τη δικαιοδοσία, γιατί αν δεν έχουμε δικαιοδοσία δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε έρευνα. Δεύτερον, όπως λέει και ο κανονισμός, μπορούμε να το κάνουμε μόνο εφόσον υπάρχουν ουσιαστικές υποψίες για απάτη. Τρίτον, επί τη βάση της αρχής ε, της επικουρικότητας μπορούμε να ξεκινήσουμε ε, μπορούμε μόνο να ξεκινήσουμε μια έρευνα αν υπάρχει προστιθέμενη αξία γι' αυτό, γιατί διαφορετικά προωθούμε τις εισερχόμενες πληροφορίες στους, στις εθνικές αρχές. Ωστόσο, Ο αριθμός των ανοιχτών δρευνών ε, αυξάνεται διαρκώς. Για τα τσιγάρα και το λαθρεμπόριο. Θα μπορούσα ταυτόχρονα να απαντήσω σε δύο μέλη, στην κυρία Γκρέσλε και στον εισηγητή. αυτόχρονα. Και πάλι με την αναδιοργάνωση, δηλαδή μόνο από 1η Δευτέρου 2012 ως τμήμα της αναδιοργάνωσης, σαφώς είμαστε μοιρασμένοι εντός της, Ένωσης, εντός ΟΛΑΦ. Ε, Έχουμε μοιράσει τις ερευνητικέ μας ε, ε, μονάδες από την εργασία πολιτικής. Για τα τσιγάρα, ας πούμε, αυτό σημαίνει ότι η προηγούμενη μονάδα υπεύθυνη για τα τσιγάρα που ταυτόχρονα ασχολείται και με την πολιτική της Όλαφε σε αυτό το τομέα, ε, διαιρέθηκε τώρα σε δύο διαφορετικές διευθύνσεις και τώρα αυτοί που ασχολούνται με τις έρευνες για τα τσιγάρα δεν κάνουν και την πολιτική και τούμπαλιν. Ε, δεν υπάρχει δηλαδή σύγχυση αυτών των δύο ρόλων. Δεύτερον, αλλά και για τις δύο αυτές τις δυνατότητες, δηλαδή πολιτική και έρευνα, έχουμε κάνει πολλά <coughs> τα τελευταία δύο χρόνια, φέτος δηλαδή και το 2011, για, όπως σας είπα, πρόγραμμα δράσης για την, το λαθρεμπόριο καπνού και προϊόντων καπνού στα ανατολικά σύνορα και τώρα για την αναβάθμιση αυτής της πρωτοβουλίας, δηλαδή ανακοίνωση μαζί με την Κομισιόν βεβαίως, γιατί ε, φτιάχνουμε μια ανακοίνωση για το λαθρεμπόριο του καπνού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι μια πολύ μεγάλη πρωτοβουλία από πλευράς της Κομισιόν και για τα κρατημέλη γιατί θέλουμε να εγκριθεί μέχρι την άνοιξη του χρόνου. Φυσικά το θέμα της, του λαθρεμπορίου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δουλεύουμε γι' αυτό με όλα τα κράτη-μέλη. Και είδαμε πολύ καλή, πολύ συνεργασία από τα κράτη-μέλη, γιατί είναι κοινό ο στόχος. Και είμαι πεπισμένος ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα συντονισμού και ταυτόχρονα προστασία των κρατών μελών. Αρκούν αυτά. Το νέο 1073 ήδη έλαβα θέση περί αυτού. Δεν μπορώ παρά να επαναλάβω αυτά που έχω ήδη πει. Ότι δηλαδή η τροποποιημένη εκδοχή του 1073 είναι σωστή, την καλωσορίζω. Δεν θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στην ε, ε, ζωή της Όλαφ, γιατί ήδη έχουμε λάβει υπόψη όλες τις βασικές αλλαγές, επίσης σε σχέση με, όχι ακριβώς, τη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων από πλευράς των ερευνών μας. Αυτό ήδη λαμβάνεται υπόψη και εφαρμόζεται τουλάχιστον από την 1η Δευτέρου 2012 με τη νέα διαδικασία έρευνας. Οπότε στην πράξη ελπίζω ότι αυτή η πρωτοβουλία, ε, η νομοθετική, θα εγκριθεί από το Κοινοβούλιο σύντομα. Έχουμε ήδη προβλέψει τι συμβαίνει στο κείμενο και δεν θα χρειαστούν σημαντικές αλλαγές. Αυτό όμως το οποίο μας προκαλεί και πρέπει να το επαναλάβω είναι ένας πολύ βασικός λόγος ανησυχίας είναι βέβαια το θέμα της, ε, του προπολογισμού και των περικοπών και πώς αυτό θα αντικατοπτριστεί στις δυνατότητες της Όλαφ για περισσότερο, όχι, όχι περισσότερο προσωπικό, αλλά τουλάχιστον να μην περικοπεί κιόλα. Μας ανησυχεί αυτό πολύ. Συνδυασμένο αντίκτυπο των νέων διαδικασιών και απαιτήσεων τη νέα νομοθεσία, συν, όπω είπα σήμερα, η τεράστια αύξηση εισερχόμενων πληροφοριών, δηλαδή η τεράστια ζήτηση με το τέταρτο στοιχείο τις περικοπές προσωπικού, καταλάβετε γιατί ανησυχούμε για το εγγύς μέλλον και θα ήθελα να σας ρωτήσω, να, το, να σας ζητήσω να μας βοηθήσετε, κύριοι Ευρωβουλευτές. Πρέπει να κλείσω, αλλά προηγουμένως να απαντήσω στην κυρία Γκρέσλε. Υπάρχει ένας μόνο, ένα μόνο νούμερο που ε, γνωρίζω και είναι στην έκθεση. για την ε, έρευνα. Είναι ακόμα ένα ρεκόρ. Ακόμα ένα ρεκόρ και ο λόγος Γι' αυτό είναι σημαντικός να είμαι λίγο πιο συγκεκριμένος. Για πρώτη φορά, όπως είπαμε, στο νηποσημείωση έχουμε συμπεριλάβει στην έρευνά μας και στη μέτρηση για το μάκρος της έρευνας όλες τις συνεχιζόμενες έρευνες και όχι μόνο αυτές που είχαν τελειώσει. Διατηρώντας λοιπόν όλες αυτές τις έρευνες σε ένα ντουλάπι και μόνο κλείνοντας τις φρέσκες έχουμε πολύ μικρή διάρκεια έτσι. και ένα νούμερο το οποίο δεν μπορεί να σταθεί ε, μόνο του. Εδώ στην έκθεση που έχετε έχουμε δει όλες τα νούμερα, όλες τις ανοιχτές κρεμμύς έρευνες και όχι μόνο αυτές που έχουν κλείσει. Γι' αυτό το λόγο η μέση διάρκεια είναι κάπως μακρύτερη. Μπορώ να σας πω ότι έχει μειωθεί σημαντικά. Αλλά βέβαια δεν μπορεί να έχει και περισσότερη και καλύτερη και περισσότερη επιλογή εισερχόμενων πληροφοριών με λιγότερο κόσμο. Ακόμα προσπαθούμε μέχρι τώρα τα καταφέρνουμε, το χειριζόμαστε το θέμα. Από ό,τι κατάλαβα ο κύριος Σκυλακάκης δεν ζήτησε απάντηση, απάντηση. Οπότε Κατάλαβα ότι, ότι η ερώτησή σας δεν αφορά άμεσα την έκθεση, αλλά είμαι στη διάθεσή σας ε, για να απαντήσω για σε ό,τι επιθυμείτε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κέσλερ. Αν ε, η συγητή είναι ικανοποιημένος, ολοκληρώνουμε έτσι τη συζήτηση της ε, του, του σημείου 3 της ημερήσιας διάταξης και προχωράμε στις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες ε, η γραμματεία μου είπε ότι το 7 θα είναι πρώτο, γιατί η κυρία της πρέπει να φύγει σύντομα. Αν είστε λοιπόν έτοιμοι, προτείνω να προχωρήσουμε με το σχέδιο έκθεσης της κυρίας Ρωτής για τη μεταρρύθμιση της κοινή οργάνωσης αγοράς ίνου. Τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά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 Προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 9. Ψηφίσατε όλοι. πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10 έχει αποσυρθεί. Τροπολογία 11. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ποιο είναι υπέρ κατά. Προτείνω να Κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Of amendment 11 in favor against abstentions adopted. Για το 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, απορρίπτεται, με συγχωρείτε. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ελεγχός ηλεκτρονικός. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Διαδικαστικό Γερμπράντι. Μπορούμε να ψηφίσουμε χωριστά την παράγραφο 17 παρακαλώ. Όχι μόνο για την τροπολογία πι της παραγράφου, αλλά για την παράγραφο την ίδια. Αν συμφωνεί ο εισηγητής ή η εισηγητρία. Δεν έχω πρόβλημα, αλλά η παράγραφος 17 Έχει μόνο μία δυνατότητα ψήφισης. Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Κύριε Γερμπράντη, μπορείτε να εξηγήσετε λίγο. Ναι, έχουμε την παράγραφο 17 και έχουμε και μία τροπολογία που αφορά την παράγραφο 17, που είναι και η τροπολογία 17. Έχει και τον αριθμό 17, η ίδια η τροπολογία, ίσως εκεί τη σύγχυση. Εγώ θα ήθελα να ψηφίσουμε χωριστά για την αρχική παράγραφο πριν ψηφίσουμε επί της τροπολογίας. Εγώ προχω, ε, προ, προτιμώ να γίνει αυτό που έχουμε προτείνει. Δηλαδή, να, μόνο το κομμάτι 17 έχει διάφορα εδάφια και η 17 όχι. Προτιμώ να παραμείνει ως έχει. Κύριε Γκρέσλε τα δύο αυτά πρέπει να συντονίσουμε τις παραγράφους οι οποίες αλλάζουν διότι διαφορετικά θα πρέπει να προβούμε σε διαγραφή. Ε, συμφωνώ με τον ε, εισηγητή διότι εφόσον υπάρχει ε, κατάπτωση της τροπολογίας ε, σημαίνει ότι με τροπολογία υποκαθιστάται η παράγραφος 17 από ένα διαφορετικό κείμενο. Έχουμε ένα κατάλογο ψηφοφορίες και έτσι ακολουθούμε. Ε, ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 17. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Λίγη. Ενεκρίθη και συγχαίρω τον εισηγητή. Την εισηγήτρια. Το επόμενο θέμα είναι η έκθεσή μου σχετικά με την ε, την ε, πρόθεση δράσεως προστασίας των οικονομικών συμφερών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ε, δεύτερη σελίδα, ΚΑΤΑ ενεκρίθη. Η 32 είχε αποσυρθεί, τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6, τροπολογία 34 και 7 από κοινού τις ψηφίζουμε. 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 35 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ, αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προϋπολογισμός 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Προπολογιά 11 υπέρ κατά εποχές, Δεν είμαι βέβαια, ας το ελέγξουμε για την 11. is Εγκρίνεται. Καταπίπτει λοιπόν 10 την προϋπολογισμού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 41 υπέρ κατά... Για να κάνουμε έναν ηλεκτρονικό έλεγχο στη 41. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 42 έχει αποσυρθεί. 43. Περ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προπολογισμού 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 προπολογισμού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προπολογισμού 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 κατά πίπτη, ε, προϋπολογισμό 14 υπέρ κατά. Ας κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για την ε, τροπολογία 14 της Επιτροπής Προπολογισμού. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 47 υπέρ. Δεν βλέπω χέρια να σηκώνονται. Υπέρ ποιοι είναι. Κατά απόχέ εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 15 προπολογισμό εγκρίνεται. Υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται. 48 έχει αποσυρθεί. Συμβιβαστική ε, α σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Ηλεκτρονικός έλεγχο. Πρώτο τμήμα τη συμβιβαστική α. Τέλος της πληροφορία. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της συμβαστικής α, υπέρ ηλεκτρονικά. Όχι, όχι, όχι, εντάξει, είναι σαφές, εγκρίθηκε. Τροπολογία 49, 49, 50 και 17 καταπίπτουν και πάμε στην προφορική των πρασίνων υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 18 προπολογισμό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 κατά πίπτη 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 προπολογισμό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 με προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 έχει αποσυρθεί. 3 προπολογισμού υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προπολογισμό 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Οι σοσιαλιστές τι είναι, υπέρ, κατά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά τότε για την ε, προ, ε, ε, τροπολογία 5 της επιτροπή Προπολογισμού. Τέλος φωτορίας. Εγκρίνεται. 6 προϋπολογισμό υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 26 έχει αποσυρθεί. 27 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 7 η προπολογισμό έχει καταπέσει 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και ε, ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Τώρα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για το σύνολο της έκθεσης όπως τροποποιήθηκε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Επόμενο σημείο τώρα. Α, συγγνώμη, η νομοθετική πρόταση πρέπει να ψηφιστεί τώρα. Ψηφίζουμε. Η πρόταση νομοθετικού ψηφίσματος, τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Επόμενο σημείο. Ναι, ευχαριστώ. Θα ήθελα μάλιστα να ευχαριστήσω όλους τους Σκεώδης για την εξαίρετη συνεργασία. Γκάιερ, Σκυλακάκης, ε, ε, Σαΐς, όπως ξέρετε θα φύγω από το Κοινοβούλιο στα τέλη του έτους και κάποιος άλλος θα αναλάβει το θέμα αυτό. Αποφασίστηκε από το ΕΛΚ η κυρία Μακοβέη θα με διαδεχθεί, οπότε θα ήθελα να ρωτήσω αν έχει κανείς αντιρρήσεις ε, να ηγηθεί εκείνη της διαπραγματευτικής ομάδας και να χρησιμοποιήσει αυτό το υιοθετημένο κείμενο ως βάση για τις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενο θέμα, έκθεση ΣΤΑΕΣ. Σχέδιο έκθεσης για την ειδική έκθεση ε, ε, 2011 για την ε, ιατροφική ασφάλεια στην υποσαχάρια Αφρική. Κύριε Σκυλακάκη, θέλετε να πείτε κάτι, ναι, αν είναι δυνατόν να... Εκτός από την τροπολογία 7 και 8, τα υπόλοιπα να τα ψηφίσουμε εν μπλοκ, γιατί νομίζω πως γίνεται. Μπορεί να γίνει. Ένα μέχρι 12 είναι οι τροπολογίες. Όχι λέτε. Okay. made an πάντων, την έκανα την προσπάθεια. Ένα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δύο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρία υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Έλεγχος ηλεκτρονικός στις τρία. Τέλος ψηφοφορίας. απορρίπτεται. 4 υπέρ με την προφορική. Ψηφίζουμε για τροπολογία 4 με την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για τροπολογία 7. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 8 υπέρ ηλεκτρονικός έλεγχος. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εάν θέλετε να ελέγξουμε, ας ελέγξουμε. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 9. Υπε... τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Μέχρι και 12 unblock. 10. Υπέρ ποιοι είναι. Αποχές εγκρίνονται. Και τώρα Ψηφίζουμε για τις τροπολογίες της Επιτροπής Ανάπτυξης. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε. 5 της Επιτροπής Ανάπτυξης υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την 5 τέλος της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Οι 6 και 7 καλύπτονται, 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε το σύνολο της έκθεσης όπως τροποποιήθηκε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια, κύριε Στάις. Σημείο 6. Οντι. Θέλετε το λόγο? Ναι, Πρόεδρε. Για τις τροπολογίες ΑΦΕΤ θα πρότεινα μετά από διάφορες διαβουλεύσεις να τις ψηφίσουμε unblock εκτός από την 7. Ε, Για δεν υπάρχει αντίρρηση βέβαια. So, is there any objections to taking amendment from one to... Υπάρχει καμιά αντίρρηση να δούμε από κοινού την στροπολογίες ε, 1 μέχρι 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Την 1 τώρα υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Ψηφίζουμε τώρα για το σχέδιο έξεσης όπως οτροποποιήθηκε. τροποποιήθηκε. Τέλος ψηφοφορίας. That is adopted. Congratulations to... Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Και έτσι ολοκληρώσαμε τις ηλεκτρονικές μας ψηφοφορίες. Και συνεχίζουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας μας διάταξης που είναι το υπερφών 8, αντιπροσωπεία της, αποστολής, της ε, περιτροπής μας στους λιμένες του Ρότερταμ και της Αμβέρσας. 19 και 20 Σεπτεμβρίου έγινε η επίσκεψη. Η έκθεση έχει σταλεί στους ευρωβουλευτές για σχόλια και προτάσεις και σήμερα έχω τη χαρά να σας παρουσιάσω αυτή την έκθεση. Ε, θα περιμένω ένα-δύο λεπτά για αυτούς που δεν ενδιαφέρονται για την έκθεση σχετικά με το λιμάνι του Άμστερνταμ και της Αμβέρσας να έχουν εγκαταλείψει την αίθουσα και μετά θα ξεκινήσω.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 θα ήθελα να ευχαριστήσω αυτούς οι οργάνωσαν αυτές τις επισκέψεις και ε, ε, μας έδωσαν τις πληροφορίες όπως και τους συναδέλφους που συμμετείχαν διότι ε, ουσιαστικά αποτελούν το 13% των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και η Αμβέρσα και το Ρότερνταμ είναι τα δύο μεγαλύτερα λιμάνια και γι' αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον για μας να διαπιστώσουμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα δικαιώματά της προστατεύονται. Καταρχήν όπως γνωρίζετε πήγαμε για να δούμε πώς γίνεται και ο έλεγχος των γράφων αλλά συγχρόνως και ο φυσικός έλεγχος πώς εφαρμόζεται η νομοθεσία στην πρακτική και να διαπιστώσουμε και τις ε, αδυναμίες ε, της ε, παραδοσιακής απόδοσης των ιδίων πόρων. Είχαμε στην Ολλανδία πρώτον ανταλλαγές απόψεων με τους εκπροσώπους του λιμανιού του Ρότερνταμ. Είδαμε το μεγαλύτερο σταθμό διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων. Είδαμε το πόσον ποσό των κατεσχεμένων εμπορευμάτων και διαπιστώσαμε την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ελέγχου. Ε, το βράδυ συναντήσαμε τους εκπροσώπους της ε, βιομηχανίας ε, καπνού που εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για την παραποίηση των εισαγωμένων προϊόντων καπνού και τσιγάρων. Ε, είδαμε και τον συνοριακό σταθμό ε, και στις συνεδριάσεις αυτές οι αρχές μας έδωσαν στοιχεία σχετικά με τις κατασχέσεις ναρκωτικών και τσιγάρων για την περίοδο 2010-2012 ε, και για να είμαι σύντομη θα σας πω που καταλήξαμε ως συμπεραράσματα ότι ο ανταγωνισμός δεν πρέπει να μας οδηγήσει σε μία υπερβολική απλοποίηση των συστημάτων ελέγχου και θα πρέπει να υπάρχουν τα εχέγγια ότι προστατεύονται σωστά οι ίδιοι πόροι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι ε, ποιες, ε, ε, ε, πώς είναι ο χειρισμός για τους ίδιους πόρους. Δεν θα πρέπει να κλείνει ο φάκελος εάν δεν έχει διαπιστωθεί ότι οι έμποροι έχουν συμμορφωθεί προς την νομοθεσία και οι δηλώσεις θα πρέπει να ελέγχονται καλύτερα για να μειώνονται και οι έλεγχοι. Τέλος ε, θα πρέπει να παραμείνει το θέμα αυτό προτεραιότητα διότι είδαμε ότι ε, υπήρχαν υπήρχαν πολλές κατασκέσεις και αυτό ήταν προς όφελος της υγείας των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, τέλος όσον αφορά την κατανάλωση παραποιημένων ή λαθρέων τσιγάρων είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να απασχολήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία να προβεί εις ελέγχους ε, προς ε, την πηγή ε, προελεύσεως για να μπορέσουμε να καταλύσουμε. Αυτή είναι ουσιαστικά η έκθεσή μου ε, και θέλω να ευχαριστήσω τους συμμετέχοντες στην έκθεση. Χαιρετίζω οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε να μου κάνετε ή αν υπάρχει κάτι το οποίο θέλετε να μου πείτε. Η... Υπάρχουν εκπρόσωποι της ε, ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την έκθεση αυτή η οποία αντικατοπτρίζει πολύ σωστά τις συναντήσεις με τις αρχές ε, ε, στην Αμβέρσα και στο Ρότερνταμ όπου έγινε προσπάθεια να αντιμετωπίσουν τις ε, ανησυχίες μας θεωρήσαμε ότι ήταν μια επιτυχής επιχείρηση και Πρέπει να σας πω ότι ο υπεύθυνο δεν είναι εδώ σήμερα διότι ε, ε, ε, απουσιάζει σε αποστολή και έχω ένα μόνο σχόλιο σχετικά με τα συμπεράσματά σας εις το σημείο που λέγεται ότι η έλεγχοι εξ πόστο γίνονται ε, είναι τυχαίοι. Δεν πρέπει όμως ε, να ε, είναι μόνο τυχαίοι, πρέπει να βασίζονται και σε μια ανάλυση κινδύνων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, είμαι ε, υπεύθυνος από την ε, Διεύθυνση Προπολογισμού και είμαι υπεύθυνος για την, της, τον έλεγχο των ιδίων πορών και κάνουμε μέσω της διευθύνσεώς μου τις επιθεωρήσεις στα κράτη-μέλη αλλά καταλήγω στα ίδια συμπεράσματα με τη, τα πορίσματα της αποστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε κάνει σε όλα τα κράτη-μέλη τέτοιες μελέτες και πέρυσι ε, στην διαδικασία διακίνησης και εκτελονισμού των προϊόντων είχαμε παρουσιάσει πέρυσι στα κράτη-μέλη μία έκθεση και εφέτος το Δεκέμβριο θα παρουσιάσουμε την έκθεση για τον εκτελονισμό επιτόπου ε, συμφωνούν και συνάδουν τα συμπεράσματά μας με αυτά των εκθέσεών σας και καταλήξαμε ότι οι απλοποιημένες ε, ε, τελωνιακές διαδικασίες δεν εμποδίζουν τις αρχές να προβαίνουν στους ελέγχους ε, και μπορούν βάσει αυτών των ε, στοιχείων να εστιάσουν τους ελέγχους και ε, θα χρειαστεί περισσότερη συνεργασία και εντός ε, των κρατών μελών ε, και γενικότερα σχετικά με την ε, αυτόματη ανάλυση κινδύνων την οποία εφαρμόζουμε. Ε, θεωρήσαμε ότι πρέπει να ενισχυθούν οι έλεγχοι στα κράτη-μέλη ε, για να δούμε ε, τι θα γίνει στη συνέχεια και θα πρέπει να συνδυάσουμε τις εμπορικές διευκολύνσεις με τους ελέγχους και διαπιστώνουμε ότι η εφαρμογή της νομοθεσίας δεν έχει ολοκληρωθεί και παρακολουθούμε εκ του σύγκυνηγης ε, τα πορίσματα των ε, ε, επιθεωρήσεων και στο μέλλον θα ασχοληθούμε και με τους αποτελεσματικούς ελέγχους διότι ε, έτσι ε, ε, έχουμε κάτι το οποίο είναι προς όφελος των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Εάν δεν υπάρχει, ο κύριος Μίλντερ έχει το λόγο. Ήθελα να σας πω ότι υπήρξαν ε, ορισμένες εκθέσεις στον τύπο και αντιλαμβάνομαι ότι τα σχόλια που υπήρχαν στον τύπο στη Βουλγαρία δεν αναφέρονται σε εσάς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Γκρέσλε. Με συγχωρείτε, απλώς ήθελα να σας πω ότι έχω την εντύπωση ότι δεν ε, κοιτάζουμε ε, ορισμένα θέματα και ε, εάν δεν υπάρχουν έλεγχοι καταλήγουμε στο αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που θα θέλαμε. Καλό θα ήταν λοιπόν να εξετάσουμε τι γίνεται με τους χρήστες και ξέρουμε ότι το Ρότερνταμ έχει μία ιδιάζουσα φήμη δεν πρέπει λοιπόν επουδενή λόγο εμείς να συμπράξουμε σε παρατυπίες ε, θα έπρεπε να το, να το λάβει υπόψη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί δεν είναι προσόν να υπάρξει μία μείωση των ελέγχων. Ευχαριστώ. Άλλα σχόλια. Αν όχι, σας ευχαριστώ όλους. Αυτό ολοκληρώνει την ημερήσια διάταξη για σήμερα και προχωράμε στην εδρίαση των συντονιστών.